Επομένως, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφη 3 και 4 του κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στην συνεδρίασή της της 19 Μαρτίου 2014 ε, επαλήθευσε τις εξουσίες του κυρίου Τζοβάνι Μπαρμπαγκάλο και της κυρίας Ανέτ Κεβιούς και προτείνει την επικύρωση της ε, ε, εντολής και των δύο βουλευτών ε, με έναρξη ισχύω την 11η Μαρτίου 2014 για τον κύριο Μπαγκάλο και τις 12 Μαρτίου για την κυρία Κέβιους. Σας προτείνω λοιπόν να επικυρώσετε αυτές τις εντολές. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Όχι, επομένως επικυρώνονται και συγχαίρω τους δύο συναδέλφους. Ο κύριος Μπρίσε Ορτεφέ υπέβαλε στο Προεδρείο αίτημα υπεράσπισης της βουλευτικής του ασυλίας